E λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι, επίτροπε επανερχόμεθα. Το επόμενο θέμα είναι η έκθεση του κυρίου Γκούναρ Χέκμαρκ για την πολιτική στον τομέα του ραδιοφάσματος. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Χέκμαρκ. Πρόεδρε, επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Αυτή η έκθεση ε, έχει ως στόχο να, να, να ανέβει στην πρώτη θέση η Ευρώπη. Είναι επίκαιρη λοιπόν η σημερινή μας συζήτηση. Το 50 όταν ε, ο Σούμαν ε, εισηγήθηκε την ίδρυση της κοινότητας αυτής μίλησε για το ατσάλι και το χάλιβα. Ε, τώρα ασχολούμαστε με τις νέες τεχνολογίες και τις γνώσεις. Αυτά θα έχουν την καθοριστική σημασία για το μέλλον της Ευρώπης. Με χαρά μπορώ να σας πω ότι η έκθεση που παρουσιάζουμε εδώ σήμερα προέκυψε από μια πολύ αγαστή συνεργασία με τους σκιώδεις εισηγητές, η κυρία Τράουτμαν, ο κύριος Τράουντερ, ο κύριος Τσίτσεστερ και η κυρία Λαμπέρτα υποστήριξαν αυτή την έκθεση. Χαιρόμαστε όλος ιδιαίτερος διότι σήμερα εξετάζουμε μία πρόταση χάρη στην οποία μπορεί να διατηρήσει τον ηγετικό της ρόλο η Ένωση για την κινητή τηλεφωνία, το κινητό διαδίκτυο και τις ε, σύγχρονες ε, κινητές τεχνολογίες. Πρόεδρε, κατά τη γνώμη μου, η συζήτηση που κάνουμε για τις επιμέρους προτάσεις της έκθεσης αυτής ουσιαστικά σχετίζεται με μια επιλογή. Δηλαδή, η Ευρώπη θα επιλέξει να έχει την πρωτιά ή θα αρκεστεί στην τρίτη θέση. Είναι μια απλή επιλογή, τουλάχιστον όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ. Ορισμένες φορές όταν συζητούμε σχετικά με το ποια είναι η μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο, όλοι αναφέρονται στη ΣΥΠΑ και στην Κίνα. Ε, ξεχνούμε όλοι πως η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο. Αλλά δεν έχουμε τις μεγαλύτερες αγορές. Τώρα θα εξαρτηθεί από μας τι θα γίνει στο μέλλον. Σήμερα θα συζητήσουμε εάν θα κάνουμε τις απαιτούμενες αλλαγές ώστε να ανατραπεί αυτή η τάση. Να γίνει μια ρήξη σχέση με το παρελθόν και με διαδοχικά βήματα να κατοχυρώσουμε την πρωτιά μας στις τηλεπικοινωνίες, ε, στην ανάπτυξη της ευρυζωνικής τεχνολογίας. Εγώ προσωπικά θέλω η Ευρώπη να έχει τη μεγαλύτερη δυναμικότητα και τις υψηλότερες ταχύτητες για τις ευρυζωνικές ε, συνδέσεις. Ε, γιατί τότε θα υποδεχθούμε όλες τις νέες υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν στη δική μας Ήπειρο και θα έχουν και με τη σειρά τους καθοριστική σημασία για την αναπτυξιακή πορεία της Ευρώπης. Για την επόμενη γενιά όλων αυτών των ε, μηχανημάτων ανέβρεσης, ε, Google, Yahoo, όλες αυτές οι εταιρείες ε, που έχουν βγάλει το μανιφέστο τους για την καινοτομία. Εμείς μπορούμε να υποδεχτούμε όλες αυτές τις νέες εταιρείες βέβαια και άλλες οικονομίες όπως η ΕΠΑ, ΕΕ, η Κίνα και η Ινδία θα επιδιώξουν την πρωτιά. Άρα πρώτα απ' όλα θα πρέπει να κάνουμε αυτή την επιλογή που προανέφερα σε σχέση Τώρα με τα 800 GHz και την ζώνη ραδιοφάσματος μέχρι το 2013 προτείνω να μην περιοριστούμε σε αυτό. Θέλω να είμαστε ακόμη πιο φιλόδοξοι. Ε, να απελευθερώσει 1200 MHz η Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι τα 2,5 MHz δηλαδή και, ε, από το 1,8 μέχρι το 2,5 και επίσης να εξετάσει και την απελευθέρωση της ε, συχνότητας των 7 MHz. Δεν θα μπορέσουμε στο μέλλον να πάρουμε τέτοια τέτοια απόφαση, τα 5 MHz μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε για ελεύθερη χρήση, άνευ άδειε για τι χρήσει σύντομη, ε, μικρή απόσταση μάλλον, φυσικά μιλώντα για την κινητή τηλεφωνία. Έχετε λοιπόν την πρόταση πλέον μπροστά σας και θα ήθελα να συνεχιστεί ο διάλογος και με τα κράτη-μέλη, ώστε να τους ε, ρωτήσω ακριβώς ε, αυτό. Θέλετε να είστε πρώτοι ή θα αρκεστείτε στην τρίτη θέση. Αυτή είναι η βασική ερώτηση και προσβλέπουμε ανυπομοσία στην τριτη θεση αυτη ειναι η βασικη ερωτηση και προσλεπουμε ανυπομοσια στην ψηφοφορια που θα γίνει ε, την Πέμπτη. Ευχαριστούμε. Η κυρία Κρόστορα έχει το λόγο, η αρμόδια Κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη του Κοινοβουλίου, νομίζω ότι εδώ έχουμε ε, μια προειδοποίηση η οποία μας γίνεται. Αυτό μας μεταφέρει πραγματικότητα και γι' αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω από πλευράς μου τον εισηγητή, τον κύριο Χάκμαρκ, γιατί έχει κάνει εξαιρετικά σκληρή δουλειά σε σχέση με ε, το πρόγραμμα για το ραδιοφάσμα. θα πρέπει να αποφασίσετε τι θέση θα πρέπει τελικά να πάρει η Ευρώπη γύρω από το θέμα αυτό. Όλο προς τη Δύση, όλο προς Ανατολάς, το μέσο αυτής της απόστασης, αλλά σίγουρα η Ευρώπη πρέπει να διεκδικήσει την πρώτη θέση. Αναφέρομαι σε ένα πρόγραμμα το οποίο είναι ουσιαστικά για την ψηφιακή ευρωπαϊκή οικονομία και για την κοινωνία μας στο σύνολό της. Είναι σαφές από την έκθεση που έχουμε μπροστά μας ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εμπολή συμμερίζεται την άποψη της Επιτροπής για τη σημασία μιας συντονισμένης πολιτικής στον τομέα του ραδιοφάσματος. Είναι ζωτικό να διατηρήσουμε και να βελτιώσουμε την ανταγωνιστική θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μεγιστοποιήσουμε τις κοινωνικές και πολιτιστικές επιπτώσεις μέσω της καινοτομίας υπέρ του πολίτη. Θα ήθελα επίσης να εμείνω και στον πολιτισμικό τομέα, στην πολιτισμική επίπτωση αυτής της πολιτικής. Μιλάμε για το διαδίκτυο, ένα από τα βατικά μέσα που δείχνουν περαιτέρω ε, ε, εξελίξεις και περισσότερα μέσα στην διάθεση της ευρωπαϊκής κοινωνίας. Μιας κοινωνίας της γνώσης και μιας κοινωνίας προχωρημένης πολιτισμικά. Πολύ σωστά είπατε κύριε ε, Ισηγητά, ότι έφτασε η ώρα της επιλογής. Δεν αρκούν τα καλά λόγια. Αυτό το κάναμε στο παρελθόν. Τώρα πλέον έχουμε πει τι χρειάζεται η Ευρώπη, τώρα έφτασε η ώρα να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Δεν μπορεί κανείς να επιδιώξει και να αναζητήσει την πρώτη θέση, την ηγετική θέση, εάν δεν ακολουθήσει τις επιλογές που οδηγούν σε αυτή. Σχετικά με τις πολιτιστικές πλευρές, κύριε Πρόεδρε, να μου επιτρέψετε να πω ότι κάποια πολιτιστικά στοιχεία πρέπει να υπογραμμιστούν περαιτέρω. Γνωρίζω ότι το θέμα αυτό είναι βασική ανησυχία των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Βλέπω ότι υπάρχουν δυνατότητες συνέργειας για τη χρήση του φάσματος και για την κατανομή πολιτιστικού ε, περιεχομένου και ε, για τον τομέα τον ραδιοφωνικό και για τον τομέα τον τηλεοπτικό και για το ευρύ φάσμα το οποίο θα πρέπει να αναπτυχθεί παράλληλα. Και γι' αυτό κυρία Πρόεδρε δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι εδώ η πρόσβαση στο ευρύ φάσμα δίνει δυνατότητα πρόσβαση σε πολιτιστικά προϊόντα και ε, πρέπει να καλυφθούν οι περιφέρειες οι οποίες δεν καλύπτονται από το εφήφασμα σε αυτή τη φάση. Η πρόταση όχι μόνο προστατεύει τις περιοχές αυτές αλλά διασφαλίζει ε, την μελλοντική ανάπτυξη αυτών των βασικών πολιτιστικών αλλά και οικονομικών ε, προγραμμάτων που προϋποθέτουν φυσικά και την παραγωγή πλούσιου πολιτιστικού περιεχομένου. Παραμένουν εμπόδια όπως τα προβλήματα που έχουμε με τις εναέριες επικοινωνίες και με την τηλεόραση ε, είναι ένα θέμα που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Αλλά ξέρουμε ότι δεν υπάρχουν πλέον στον τομέα αυτό σύνορα και οι ευρωπαϊκές πολιτικές θα πρέπει να τύχουν υποστήριξης και σε επίπεδο διεθνών διαπραγματεύσεων, όχι μόνο από τα κράτη-μέλη. Και χρειαζόμαστε βοήθεια για να διαπραγματευτούμε και με τις γειτονικές χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαι ήδη σε επαφή με κάποια υπουργεία και με ορισμένες χώρες μέλη γιατί ασχολούμαι με τα θέματα γειτονίας. Τώρα για το περιεχόμενο της ίδιας της έκθεσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να υποστηρίξει το περιεχόμενο με κάποιες μικρές τροποποίησεις. Μπορούμε όμως να πούμε ότι συμμεριζόμεθα πλήρως την άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφωνεί με την θέση του εισηγητή σε κάποια ιδιαίτερα σημαντικά θέματα. Η σημασία του φάσματος για την ψηφιακή ατζέντα θα διασφαλίσει στους, στους, πελά, στους πελάτες, στους πολίτες μάλλον, την πρόσβαση στο ευρύ φάσμα και δημιουργεί τις δυνατότητες και για περαιτέρω φάσμα για να καλυφθούν οι ανάγκες για σύρματη επικοινωνία στο μέλλον. να γνωρίζετε ότι και εμείς γνωρίζουμε ποιες είναι οι εξελίξεις οι τεχνολογικές που έρχονται γρήγορα. σχετικά τώρα με το ψηφιακό φάσμα των 800 σίγουρα απαιτούνται παρατάσεις των εξαιρέσεων μέχρι το 2013 εκεί είναι ο πρώτος στόχος που έχουμε αλλά πρέπει να υπάρξει μια δυνατότητα για περαιτέρω παράταση των εξαιρέσεων και μετά το 2013 κάτω από απρόβλεπτες τεχνικές συνθήκες και λόγω επίσης των προβλημάτων στην επικοινωνία που μπορεί να έχουμε με ορισμένες τρέτες χώρες. Υπάρχουν και άλλες ευρωπαϊκές πολιτικές πέραν της παρέμβασης στον τομέα της επικοινωνίας της ηλεκτρονικής. Αναφερόμαστε στη γεωργία, στις μεταφορές και εκεί υπάρχει ανάγκη για διάθεση ευρύτερου φάσματος στον τομέα της ενημέρωσης και θα πρέπει να καλύπτεται και με σωστό τρόπο ο τρόπος μάλλον που αντιμετωπίζεται η χρήση του φάσματος, του διαθέσιμου φάσματος από τους χρήστες. Υπάρχει ανάγκη, Πρόεδρε, να συντονίσουμε την προώθηση των ευρωπαϊκών πολιτικών όμως σε διεθνές επίπεδο και έτσι θα υποστηρίξουμε τα κράτη-μέλη στις διαπραγματεύσεις τους με τις χώρες εκτός της Ένωσης. Υπάρχουν και άλλα θέματα στα οποία υποστηρίζουμε την έκθεση η οποία ενισχύει τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε ορισμένες τροπολογίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να είναι λίγο πιο διαφοροποιημένη. Η παρουσίαση των στόχων και των αρχών δεν θα πρέπει να μειώσουν το ευρύ φάσμα της αποτελεσματικής χρησιμοτικότητας του φάσματος που θα πρέπει να εφαρμόζεται με τον μέγιστα ωφέλιμο τρόπο. Και ένα άλλο θέμα στο οποίο πρέπει λίγο να διαφοροποιηθούμε Κατανοώ την ανάγκη ε, ε, επαρκούς φάσματος για τα ραδιοτηλεοπτικά. Αυτό όμως δεν θα πρέπει να αποκλείει άλλους τρόπους μετάδοσης περιεχομένου. Μια άλλη διαφοροποίηση ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφορά τον ανταγωνισμό και για την θέση σε διάθεση μάλλον σε νεοεισερχόμενες επιχειρήσεις ε, ποσοτήτων φάσματος αυτό θα πρέπει να γίνει με τρόπο ο οποίος πρέπει να καθοριστεί καλύτερα και τότε δεν θα υπάρχουν διαφορές μεταξύ μας. Υπάρχουν θέματα και κάλυψης του κόστου συγκεκριμένων δραστηριοτήτων μέσω κρατικών βοηθειών. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να γίνει, αλλά δεν νομίζω ότι εδώ υπάρχουν διαφορές απόψεων μεταξύ μας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ορισμένες δυσκολίες για την αποδοχή δύο προτάσεων όμως. Η πρώτη πρόταση αφορά το φάσμα το οποίο τεχνικά έχει ήδη γίνει αντικείμενο εναρμόνισης και την υποχρέωση αδειοδότησης της χρήσης του φάσματος αυτού μέχρι το 2012. Δεν θα πρέπει να αντικατασταθεί από μια χαλαρότερη δέσμευση η οποία λέει ότι θα πρέπει το φάσμα αυτό να είναι διαθέσιμο για υπάρχοντες χρήστες πρέπει νομίζω να περάσουμε σε ε, αποτελεσματική αδειοδότηση της χρήσης του φάσματος, να κάνουμε βήματα προς τα εμπρός και όχι προς τα πίσω. Ένα άλλο θέμα στο οποίο έχουμε κάποιες δυσκολίες αφορά την πρόσβαση σε δορυφορικές υπηρεσίες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να είναι ικανή να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα του δορυφορικού φάσματος. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν τίθεται εκ νέου θέμα αδειοδότησης και θέμα διάθεσης του φάσματος αυτού με διαφορετικό τρόπο από τον προτινόμενο από, την το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα βρούμε νομίζω μία λύση. Θα ήθελα να κάνω και κάποιες καταληκτικές παρατηρήσεις. Τόσο το Κοινοβούλιο όσο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζουν ότι η έγκαιρη έγκριση της πρότασης είναι κάτι το ευκταίο δοθή της σημασίας, μάλλον του μεγέθους της δουλειάς που καλούμεθα να κάνουμε για να εφαρμόσουμε αυτό το πρόγραμμα. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε μια σαφέστατη δήλωση το ταχύτερο δυνατόν. Εμείς από πλευράς μας θα κάνουμε τα πάντα για να υποστηρίξουμε το εγχείρημα και είμαι πεπισμένη ότι το Κοινοβούλιο θα αρχίσει εγκαίρως ένα διάλογο για να καταλήξουμε σε συμφωνία. Ο χρόνος λειτουργεί εναντίον μας πιεζόμαστε από το χρόνο και πραγματικά αν επιθυμούμε μία λύση και αν δεν αν θέλουμε να καταλάβουμε την πρωτιά όπως μας πρότεινε ο κύριος Χέκμαρ στην εισήγησή του, ε, θα πρέπει να βιαστούμε και να βάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. <clears throat> Ε, τώρα το λόγο θα πάρει η κυρία Κάμερα Εβέρτ εκ μέρους της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας. Έχετε το λόγο κυρία συνάδελφη για ένα λεπτό παρακαλώ. Yeah, Μάλιστα σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, πολιτικές πρωτοβουλίες για μια συνολική ανάπτυξη ταχύτερων συνδέσεων με το διαδίκτυο πρέπει να χαιρετιστούν. Όμως οι συχνότητες είναι περιορισμένο αγαθό και κυρίως δημόσιο αγαθό. Γιατί η Επιτροπή Πολιτισμού ήταν κύριο αίτημα να καταστεί σαφές ότι οι συχνότητες πρέπει να χρησιμοποιούνται για πολυσχηδή, πολυσχηδές έργο στον πολιτιστικό τομέα δώσαμε ιδιαίτερη σημασία το πακέτο μέτρων για τις τηλεπικοινωνίες ε, πρέπει να ε, μην άρει αυτή την προοπτική και μάλιστα από την πίσω πόρτα και ιδιαίτερα να υπάρχει η διασφάλιση για τον πλουραλισμό των μέσων ενημέρωσης στην Ευρώπη και πρέπει έτσι να διασφαλιστεί ότι το κύριο έργο αυτό θα διασφαλίζεται και στο μέλλον. Γι' αυτό η Επιτροπή Πολιτισμού πρότεινε το 790 στη συχνότητα να μην ανοιχθεί αυτή τη στιγμή. Δυστυχώ δεν ακολούθησε η Επιτροπή βιομηχανία σε αρκε... με αρκετές αφαρμές αναφέρεται ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη συγκεκριμένα ε, συμφέροντα, όμως η Επιτροπή Πολιτισμού θα έλπιζε να είχαν ληφθεί υπόψη οι τοποθετήσεις της. Για τις συχνότητες πρέπει να υπάρχουν σαφείς ε, κανόνες ε, για, τις... για τα θέματα και του θεάτρου και της αναμετάδοσης τέτοιων παραστάσεων ή εκδηλώσεων και σε σχέση και με τη νέα τεχνολογία. Καλούμαστε όλοι εδώ να λάβουμε υπόψη την αντιστάθμιση των συμφερόντων με τον πιο ισόρροπο τρόπο υπέρ των συμφερόντων όλων. Ευχαριστώ. Το πολύ. Τώρα το λόγο θα πάρουν εκπρόσωποι των πολιτικών ομάδων για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, κυρία Δεκαστή Ιωβέρα, για δύο λεπτά παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ επίσης για την παρέμβασή σας, Επίτροπε. Θα ήθελα να ξεκινήσω συγχαίροντας τον συνάδελφο κύριο Η συγητή αυτή τη έκθεση. Η δουλειά του είναι εξαιρετική και πέρα από εξαιρετική έχει ένα πολύ μεγάλο όραμα για το μέλλον και αυτό είναι ιδιαίτερα επενέσιμο. Επίση, επιτρέψτε μου να συγχαρώ όπω το έκανε ο κύριος Έκμαρ όλους τους κοιόδης εισηγητέ. και το αποτέλεσμα του έργου ήταν η ομόφωνη υποστήριξη αυτή τη έκθεση. ομόφωνη υποστήριξη στην Επιτροπή βιομηχανία αυτή τη έκθεση. Φυσικά βρισκόμαστε μπροστά σε, ένα, σε μια έκθεση που έχει ένα στόχο. Ο στόχο είναι πώ θα βελτιωθεί η δυνατότητα, η ανταγωνιστική δυνατότητα τη Ευρωπαϊκή οικονομία σε ένα παγκοσμιοποιημένο πλαίσιο. Αυτό είναι κύριο στόχος υπό τον οποίο ε, συντάχθηκε αυτή η έκθεση και είναι σωστή αυτή η προσέγγιση θα έλεγα. Δεν θα επισέθω σε λεπτομέρειες. Θα ήθελα να επικεντρωθώ περισσότερο σε δύο άλλες πτυχές που θεωρώ ότι έχουν θεμελιώδη σημασία. Πρώτα απ' όλα βρισκόμαστε σε μια κατάσταση και αυτή η έκθεση το προτείνει όπου το ευρύ φάσμα και η κατανομή συχνοτήτων για τα 800 MHz και για τις ε, δυνατότητες που διανοίγονται θα είναι πραγματικότητα στην Ευρώπη. Πρέπει να σκεφτούμε για το μέλλον τι θα γίνει. Έχουμε υπόψη τη συχνότητα 700 MHz που έχει μια εξαιρετική δυνατότητα, ένα εξαιρετικό δυναμικό και για τα κινητά και την ανάπτυξη της κινητής ε, επικοινωνίας. Σε αυτό το πεδίο πρέπει να λάβουμε υπόψη επίσης και να αξιολογήσουμε θετικά τις προτάσεις που διατυπώνονται από την έκθεση. Δεν πρόκειται για ένα θέμα ε, ίσονος σημασίας. Πρέπει να δούμε ότι 3% είναι του ΑΕΠ ε, η συνεισφορά των τηλεπικοινωνιών και αυτή είναι η αρχή μόνο, το πρώτο βήμα. Θέλω να αναφερθώ στην ανάπτυξη, γεωμετρική ανάπτυξη των βίντεο και των οπτικοακουστικών καθώς επίσης και της τηλεπικοινωνία μεταξύ των διαφορετικών ατόμων, θεσμών ή επιχειρήσεων. Αυτή τη στιγμή το βίντεο έχει 40% όσον αφορά τις διεθνείς επικοινωνίες και αυτό είναι μόνο το πρώτο βήμα, η επιχειρησεων αυτη τη στιγμη το βιντεο εχει 40 οσον αφορα τις διεθνεις επικοινωνίε. και αυτο ειναι μονο το πρωτο βημα η αρχη Για το 2014 θα είναι 91% της τελικής επικοινωνίας των χρηστών. Προς αυτή την κατεύθυνση η έκθεση τίθεται ενώπιον ενός οράματος για το μέλλον και γι' αυτό πρέπει να υποστηριχθεί. Ευχαριστώ. Τώρα για την ομάδα Σοσιαλιστών Δημοκρατών, η κυρία Τχοτμό, για τρία λεπτά παρακαλώ. Euh, Ευχαριστώ Πρόεδρε, Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Στην, σε πρώτη ανάγνωση καλούμεθα να αποφανθούμε για αυτό το πρόγραμμα πολιτικής ραδιοφάσματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που υποστήριξε και μετέτρεψε τελικά αυτή την πρόταση που γεννήθηκε στις συζητήσεις που είχαμε για το πακέτο τηλεπικοινωνιών. Χαιρετίζω τον εισηγητή, τον κύριο Χέκμαν και τους λοιπούς και τους εισηγητές. Όλοι εργάστηκαν με ικανοποιητικό τρόπο και αυτή η έκθεση είναι εξαιρετικά τεχνική, αλλά δεν περιορίζεται αυτό. Υπάρχουν και βασικές πολιτικές προκλήσεις που ενέχει η ίδια η έκθεση. Ε, τώρα, τι διαπιστώνω εγώ, το Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπω ήταν αναμενόμενο, κάνουν την ίδια διαπίστωση, αλλά έχουν διαφορετικέ φιλοδοξίε. Ε, ε, ε, είναι διασυνοριακό το αγαθό του ραδιοφάσματο και νομίζω ότι όλοι συμφωνούν επ' αυτού. Αλλά για τι λύσει όμω υπάρχει κάποιε διαστάσει απόψεων σε σχέση με τι αναλλακτικέ λύσει για το μέλλον. Υπάρχει διαφορά απόψεων με τα κράτη-μέλη που ιστορικώ πόσο φέρουν μία ευθύνη για λόγου κυριαρχία ε, παρότι ε, η λύση στην οποία κατέληξε ο συγητής ε, δεν ε, συνάδει 100% με τις δικές μου προτιμήσεις. Παρόλα αυτά υποστηρίζω αυτή την ευρύτερη προσέγγιση, δηλαδή για μια καλύτερη διαχείριση των ραδιοφάσματος που θα ανταποκρίνεται στις κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες των λαών της Ευρώπης. Αυτό νομίζω χαρακτηρίζει και διαπνέει τη θέση του Κοινοβουλίου. Σας παραπέμπω στην έκθεση πρωτοβουλία της συναδέλφου Τόγια και στις προτάσεις των οποίων υπεραμήθηκα εγώ η ίδια για το πακέτο για την πολιτική ραδιοφάσματος, η πολιτική μου ομάδα και εγώ η ίδια επιμείναμε για τις τροπολογίες μας, ε, διότι θελήσαμε να θεσπίσουμε με μεγαλύτερη διαφάνεια ε, και καλύτερη γνώση επίσης επιθυμούμε για την τωρινή διαχείριση του ραδιοφάσματος. Επίσης υπάρχει αυξανόμενη ζήτηση για ραδιοσυχνότητες ε, από τις νέες τεχνολογίες, από την κινητή τηλεφωνία πιο συγκεκριμένα και υπάρχει ζήτηση για πιο ποιοτικέ υπηρεσίε και νομίζω ότι χρειάζεται μεταρρύθμιση τη όλη πολιτική μα για να ανταποκριθούμε σε αυτέ τι απαιτήσει. Τώρα δεν πρέπει όμω για να καλύψουμε το ψηφιακό χάσμα να χρησιμοποιήσουμε ω μοχλό το ραδιοφάσμα και να εξυπηρετήσουμε τα συμφέροντα ε, των μεγάλων επιχειρήσεων καθώ και των επιχειρήσεων που τώρα ε, ξεκινούν. Θα ήθελα κλείνοντα να σα πω κάποια πράγματα για το επόμενο στάδιο. Το είπατε κι εσεί εξάλλου. Εξ αρχή ήταν σαφέ ότι δεν δεν πρόκειται να καταλήξουμε συμφωνία στην πρώτη ανάγνωση, αλλά οπωσδήποτε θα πρέπει να καταλήξουμε μέχρι το πέρα του ενιστότο έτου σε συμφωνία. Αυτό θα έχει καθαριστική σημασία για το περιμένουν από εμά οι καταναλωτέ. Είναι απαραίτητο για να αναπτυχθεί το διαδίκτυο, όποιε και είναι οι υποδομέ που χρησιμοποιούμε. Και είναι απαραίτητο επίση γιατί πρέπει να ανακάμψει οικονομικό πώ η Ευρώπη χάρη σε αυτό το πολύτιμο αγαθό. Σα ευχαριστώ πολύ κυρία Τρότμου. Τώρα για την ομάδα ε, Συμμαχία Φιλελευθέρων, ο κύριος Ρόχτε για δυόμιση λεπτά παρακαλώ. Thank Σας ευχαριστούμε. Καλύτερες και λιγότερο δαπανηρές επικοινωνίες ε, μέσω της ε, χρήσης ασματός ε, μέχρι το 2020 αυτό είναι μια φιλόδοξη πολιτική, με φιλόδοξους στόχους πρέπει να πω και την υποστηρίζω απόλυτα αυτή την προσέγγιση. Αλλά ας το ομολογήσουμε, δεν θα είναι καθόλου εύκολο. Παρ' όλα αυτά, πιστεύω ότι με την πρώτη ανάγνωση και τη θέση του Κοινοβουλίου θα είμαστε σε θέση να κάνουμε ένα μεγάλο πρώτο βήμα προς αυτόν τον στόχο. Και ας είναι σαφές για όλους, ευρύ φάσμα για όλους. Δεν είναι μόνο η διασφάλιση του καθένα ε, θα μπορεί να ε, συμμετέχει. Είναι η συμμετοχή της ε, Ευρώπης στην παγκόσμια οικονομία ως οικονομία που θα βασίζεται στη γνώση. Αν καταφέρουμε να διασυνδέσουμε 500 εκατομμύρια πολίτες, τους δικούς μας πολίτες, οι πολίτες αυτές και οι επιχειρήσεις θα μπορέσουν να δρέψουν όλου όλους τους καρπούς της ψηφιακής οικονομίας. Ιδιαίτερα δύο πράγματα πρέπει να αλλάξουν για την Ευρώπη για να μπορέσει να φτάσει σε αυτό το στόχο. Πρώτα απ' όλα χρειαζόμαστε μια καλώς λειτουργούσα πολιτική που θα είναι υπέρ του ανταγωνισμού στις τηλεπικοινωνίες στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Γι' αυτό εισαγάγαμε κανονισμούς ε, για τον ανταγωνισμό. Τα κράτη-μέλη δεν θα έπρεπε να επιτρέπεται να ε, κατανείμουν συγκεκριμένες συχνότητες παίκτες που θα συμμετέχουν στην αγορά αν κάτι τέτοιο θα μείωνε ή θα στρέβλωνε τον ανταγωνισμό της στην αγορά. Δεύτερον, χρειάζεται μια πιο αποτελεσματική κατανομή φασμάτων και μια κατανομή που θα αντανακλά τις ε, διαφορετικές ανάγκες και τις χρήσεις ε, του ραδιοφάσματος και γι' αυτό δημιουργούμε αυτό το πλαίσιο προγράμματος όχι μόνο για την απελευθέρωση της συχνότητας των 800 MHz αλλά για να μπορέσουμε και μέχρι, το 1200, ε, μέχρι τα 1200 MHz να εκμεταλλευτούμε τις δυνατότητες στο μέλλον. Θέλω να ολοκληρώσω ευχαριστώντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, <clears throat> την Επίτροπο, τον εισηγητή και τους ε, ε, συναδέφος για μια πάρα πολύ καλή συνεργασία. Χωρίς αυτή την καλή συνεργασία αυτό το επίπεδο φιλοδοξίας δεν θα μπορούσε να έχει επιτευχθεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ρόχτε. Τώρα ο κύριος Τσίτσεστερ για την ομάδα συντηρητικών μεταρρυθμιστών για δύο λεπτά παρακαλώ. Thank you. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την Επίτροπο. Να συγχαρώ καταρχάς τον κύριο Χακμάρκ έκανε μια πολύ ε, θα έλεγα ικανή παρουσίαση και νομίζω ότι γι' αυτό πέτυχε και ένα υψηλό επίπεδο συνένεσης και εδώ συμφωνώ με τους προηγούμενους ομιλητές που τον συνεχάρισαν και αυτοί. Υποστηρίζω την επιθυμία του να νομοθετήσουμε με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε η Ευρώπη να ανταποκριθεί στις τεχνολογικές προκλήσεις στο συγκεκριμένο τομέα και να διατηρήσει μια ηγετική θέση στον κόσμο. Μιλάμε για προχωρημένη τεχνολογία. Το κομβικό σημείο εδώ είναι να πετύχουμε την απαιτούμενη ισορροπία ανάμεσα στα διαφορετικά συμφέροντα τους εκπομπής της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας, τους διαχειριστές του ευρεοσφάσματος φάσματος και φυσικά ε, τους στρατιωτικούς και τις υπηρεσίες πρώτης βοήθειας. Εδώ θα ήθελα να προειδοποιήσω ότι πρέπει να σεβαστούμε ε, την επικουρικότητα και τις εθνικές αρμοδιότητες στο συγκεκριμένο τομέα. Να προσπαθήσουμε να νομοθετήσουμε στον συγκεκριμένο τομέα είναι κάτι το πάρα πολύ δύσκολο γιατί οι τεχνολογίες οι οποίες εμπλέκονται αλλάζουν εκ των προτέρων με τέτοιες ταχύτητες και τόσο συχνά που πάντα εμείς ερχόμεθα εκ των υστέρων να προλάβουμε και δεν νομοθετούμε από πριν όλα αυτά όμως θα πρέπει να δράσουμε με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να ανοίξουμε τον δρόμο στις νέες τεχνολογίες για τη σωστή εκμετάλλευση και ε, χρήση του φάσματος. Νομίζω ότι η έκθεση αυτή ε, αυτό ακριβώς στοχεύει. Δύο λεπτά από την ομάδα των ε, Πρασίνων. Merci Madame la Présidente, je voudrais... Euh, το Πρόεδρε. Θα ήθελα να συνεχίσω αντιδρώντας αυτό που ακούστηκαν. Η Κατρίν Τροθμάν είπε ότι πολύ συχνά μας λένε ότι το ραδιοηλεκτρικό φάσμα είναι κάτι το σπάνιο. Και είναι ένα κοινό αγαθό βασικά. Κανένας δεν θεωρείται ότι είναι αυστηρά μόνος ιδιοκτήτης. Κανένας εμπλεκόμενος δεν μπορεί να υποκριθεί ότι έχει εκ των προτέρων και εκτιμένα δικαιώματα για το φάσμα. Αυτό είναι κάτι το οποίο ε, ξεκαθαρίζεται από την έκθεση αυτή. Πρόκειται για ένα κοινό αγαθό, για ένα σπάνιο αγαθό συμφωνούμε και θα πρέπει να κατανοήσουμε ποια είναι η σωστή του χρήση. Και γι' αυτό γίνεται αυτή η πλήρης ε, ε, και σε έκταση εξέταση του θέματος του φάσματος από το σύνολο των εμπλεκομένων, όπως και αυτών που υπογράμμισε ο Τζάιλς, δηλαδή τις υπηρεσίες πρώτης βοήθειας, όπως και τους στρατιωτικούς να δούμε τι χρήσης γίνεται αυτού του σπανίου αγαθού σήμερα γιατί θεωρούμε ότι δεν είναι η βέλτιστη δυνατή. Απαιτείται μια διαφανής διαδικασία για την κατανομή αυτού του σπανίου αγαθού αλλά και δυναμική ταυτόχρονα έτσι ώστε να αποφύγουμε στο μέλλον να δημιουργηθούν εκ νέου νοοτροπίες εκτιμένων. Θα πρέπει επίσης να προσέξουμε στην αρχή κατανομής και θέση σε διαγωνισμό, διάθεσης μέσω διαγωνισμών του φάσματος, γιατί όλες οι χρήσεις δεν είναι εμπορικές και δεν οδηγούν στην πρόσθεση κέρδους. Φυσικά και υπάρχει η εμπορική διάσταση, αλλά και η χρήση από την κοινή ωφέλεια, από την προστασία του πολίτη για στρατιωτικούς λόγους κτλ. Αν εφαρμόσουμε μια αγοραία λογική, αυστηρά, τότε σε αυτή την περίπτωση θα δώσουμε υπερβολικά δικαιώματα σε ορισμένους εταίρους της αγοράς, οι οποίοι από το μέγεθός τους στην ουσία θα οδηγήσουν ε, τεράστιες στρεβλώσεις στην αγορά και οι μικροί πρωταγωνιστές συμμετέχοντες δεν θα έχουν την δυνατότητα δραστηριοποίησης. Να πω επίσης ότι η συνεχώς εκτατική ε, χρήση του ραδιοηλεκτρικού φάσματος είναι κάτι το οποίο έχει ιατρικές συνέπειες. Δεν είναι το θέμα μας βέβαια, αλλά οι πολίτες μας ανισχούν γι' αυτό και δεν πρέπει να το αγνοούμε. Λοιπόν, για δύο λεπτά θα πάρει το λόγο η κυρία Φερχέγεν. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε Κρούς, για τις συχνότητες φάσματος πρόκειται για ένα πολύτιμο αγαθό, περιορισμένο αγαθό, που με ιδιαίτερη σύνεση, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις κοινωνικές πτυχές, πρέπει να διαχειριζόμαστε. Γι' αυτό το ε, Frequency Program έχει ιδιαίτερη σημασία. Πρέπει να λάβουμε υπόψη ε, οικονομικά, κοινωνικά, πολιτισμικά στοιχεία που πρέπει να χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά. Γι' αυτό για όλη τη συχνότητα πρέπει να χρησιμοποιούμε τις δυνατότητες για να είμαστε το δυνατόν πιο αποτελεσματικοί. Βάσει της πολιτικής υψηλής πρέπει να είναι το πακέτο μέτρων τηλεπικοινωνίας που εγκρίθηκε πέρσι διότι η διαχείριση των τηλεπικοινωνιακών από την Ευρωπαϊκή Ένωση και, τον, και από τα κράτη-μέλη πρέπει να ανταποκρινόμαστε στις ίδιες απαιτήσει με τον ίδιο τρόπο, με κοινό τρόπο. Πρέπει να ληφθεί υπόψη αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπό αυτό το πρίσμα θέλω να αναφέρω ότι η χρήση των ε, ψηφιακών ε, μέχρι σήμερα σε περιορισμένο βαθμό έχει προχωρήσει. Ένα άνοιγμα του φάσματος κάτω από τα 800 MHz πρέπει να γίνει λαμβάνοντας υπόψη ε, την πείρα που έχουμε συλλέξει σε αυτόν τον τομέα. Πολλά τεχνικά θέματα δεν έχουν καθοριστικά ακόμα επιληθεί και το θέμα της ε, ε, επικάλυψης συχνοτήτων και των παρασίτων των ε, προβλημάτων στις, στην χρήση του φάσματος δεν έχουν όλα τα προβλήματα ικανοποιητικά επιληθεί μέχρι σήμερα. Στην κατανομή του φάσματος πρέπει τα διαφορετικά συμφέροντα με υπεύθυνο τρόπο να αντισταθμιστούν και να εξισορροπηθούν. Λαμβάνοντας υπόψη και την κινητή επικοινωνία, τηλεπικοινωνία που πρέπει να διασφαλιστεί προς όφελος των πολιτών. Όμως ε, και ένα άνοιγμα των δημόσιων ε, ε, ραδιοφωνικών σταθμών και ιδιωτικών σταθμών πρέπει να επιτευχθεί. Πρέπει να αναπτύξουμε την Ευρώπη σε σχέση με την ψηφιακή τεχνολογία, σε σχέση με το μέλλον και την πολυπολιτισμικότητα. Ευχαριστώ. Τώρα για ένα λεπτό η κυρία Ριέρα Μαντουρέλ θα πάρει το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, Σίγουρα σήμερα πρέπει να εκφράσουμε την ικανοποίησή μας για τη διεξαγωγή αυτής της συζήτησης. Πολύ συχνά, υπερβολικά συχνά ακούσαμε ότι η χρήση του φάσματος είναι τεχνικού λέει χαρακτήρα και αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών. Σήμερα, χάρη στο σθένος αυτού του Ευρωκοινοβουλίου κατά την διαπραγμάτευση του πακέτου τηλεπικοινωνίας που με εξαιρετικό τρόπο η κυρία Κατρίν Τρότμαν είχε διεξαγάγει, ο ψηφιακός τομέας τοποθετείται εκεί που πρέπει να τοποθετηθεί, στον πολιτικό τομέα, στην σφαίρα την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι περιορισμένο το ε, αγαθό αυτό και αυτό διασφαλίζει την πρόσθετη αξία ε, που πρέπει να δώσουμε σε αυτό το αγαθό ως ε, συνομοθέτες. Δεν πρέπει να υπάρξει μετοπική αντιπαράθεση μεταξύ των διαφορετικών χρήσεων του φάσματος. Η αδιάκοπη τεχνολογική πρόοδος κάθε φορά οδηγεί στο να μπορούμε να διαθέσουμε και να μεταδώσουμε περισσότερα στοιχεία με μικρότερες ε, παρεμβολές. Μέσα σε αυτή τη δυναμική ανάπτυξη σε σχέση με την ανάπτυξη της τεχνολογίας πρέπει να βρούμε τη δυνατότητα να ανταποκριθούμε στα διαφορετικά συμφέροντα των διαφορετικών χρηστών λαμβάνοντας υπόψη την εκμετάλλευση αυτού του ε, σπάνιου αγαθού. Δεν πρέπει να υπάρξουν κερδισμένοι και χαμένοι αλλά να δεσμευτούμε όλοι σε μια βελτίωση των πραγμάτων, διαρκή βελτίωση που θα προσανατολίζεται κυρίως ε, στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κυρία συνάδελφε. Ξεπεράσετε κατά πολύ το χρόνο ομιλία και σας παρακαλώ πολύ δεν μου είναι ευχάριστο να σας διακόπτω. Σεβαστείτε το χρόνο που έχετε στη διάθεσή σας γιατί γίνεται ει βάρος των συναδέλφων. Ο κύριος Οντί για δύο λεπτά. minutes, monsieur Ευχαριστώ Πρόεδρε και ε, Αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, κυρία Κρό, ε, αγαπητοί συγητά, αγαπητοί συνάδελφοι. Πρώτα απ' όλα να συγχαρώ τον συγητή, τον κύριο Χόικμαν, είναι εξαιρετική η έκθεσή του και δείχνει ανοιχτό πνεύμα. Το έδειξε εξάλλου καθ' όλη τη διάρκεια της συζήτησης και καταρχήν συμφωνεί η πρόταση με την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δηλαδή από 1η 2013 θα απελευθερωθεί η ζώνη των 800 MHz, θα χρησιμοποιηθεί για την ψηφιακή τηλεόραση και θα κατά αργηθεί η αναλογική ραδιοφωνική μετάδοση σε αυτή την ζώνη. Αυτή η χρήση από την ε, τηλεόραση απαιτεί ε, ένα μια μεγάλη ζώνη συχνοτήτων από το ραδιοφάσμα ε, ούτως ώστε να καλυφθούν οι απαιτήσει των κτηρίων και αυτές οι συχνότητες είναι γνωστές ως οι χρηστές, χρυσές συχνότητες. Μέχρι το 2015 θα πρέπει να αποφασιστούν στρατηγικά ζητήματα για την Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς την διαχείριση του ραδιοελεκτρικού φάσματος. Θα ήθελα να τονίσω δύο βασικά κατά τη γνώμη μου σημεία μέσα στην έκθεση. Αγαπητέ Γκούναρ, κύριε Επίτροπε, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να γίνει μια απογραφή που προτείνει το άρθρο 8, δηλαδή είναι ε, ε, προτιμότερο να κάνουν την απογραφή πρώτα οι εμπειρογνώμονε ε, για τι εφιστάμενε συχνότητε πριν αρχίσουμε να διαρευνούμε τη δυνατότητα χρήση εναρμονισμένων συχνοτήτων. Τώρα, ε, εάν θα πρέ... μπορεί να χρειαστεί για τις ασύρματες επικοινωνίες να βασιστούμε σε αυτήν την απογραφή. Δεν μπορούμε να προδικάσουμε βέβαια το αποτέλεσμα. Πρέπει οι προγνώμονες να επιληφθούν τους ζητήμους και να εξετάσουν τη χρήση ε, κάθε υποζώνης ε, συχνοτήτων. Δεύτερο θέμα, η χρήση των ζωνών που χρησιμοποιούνται προς το παρόν για στρατιωτικούς σκοπούς. Είναι αδιαμφισβήτητο ότι αρμοδιότητα καμία δεν έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την στρατιωτική χρήση ζωνών του ραδιοφάσματος οπότε συμφωνώ με την τροποποίηση του άρθρου 7.3 ε, και τη σχετική τροπολογία που αναφέρεται στις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για την ε, διαχείριση του ραδιοφάσμου και που παγορεύει την παρέμβαση της Επιτροπής σε στρατητικούς σκοπούς χρήσης συχνοτήτων. Ευχαριστώ πολύ, Madam Commissioner. Decizia discutată Η συζήτηση σήμερα καθορίζει το πρώτο πρόγραμμα για το ραδιοφάσμα. Η εναρμόνιση των τρόπων χρήσης του ραδιοφάσματος έτσι ώστε να διασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Στην ουσία το πρόγραμμα θα αδειοδοτεί τις δυνατότητες χρήσης του φάσματος και θα μεγιστοποιεί την ελαστικότητα χρήσης του καθιστώντας τη χρήση αυτή μέσω του συστήματος αδειοδότησης πιο αποτελεσματική, αποτρέποντας στρεβλώσεις και αποτρέποντας επίσης τεχνικές, ε, ε, τεχνικά προβλήματα στο μέλλον. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μαζί με τα κράτη-μέλη θα φτιάξουν ένα κατάλογο των υπαρχουσών χρήσεων και των δυνητικών χρήσεων στο μέλλον, ιδιαίτερα στα πλαίσια της, ε, του φάσματος από 300 MHz μέχρι 3 GHz. Νομίζω ότι όλοι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στις υποδομές αυτού με ταχύτητες 30 Mbit ανά δευτερόλεπτο το 2020. Αυτό θα διασφαλίσει δυνατότητες και για τον εμπορικό τομέα και για τις δημόσιες υπηρεσίες μέσω της σωστής χρήσης του ευρεοσφάσματος. Ζητάμε επίσης νέοι εξοπλισμοί να είναι διαθέσιμοι για τους καταναλωτές τάχιστα έτσι ώστε το πέρασμα στην ψηφιακή τεχνολογία και η χρήση ε, του ε, ψηφιακού κεκτημένου να είναι κάτι το εύχριστο για τον καταναλωτή θα πρέπει να βελτιωθεί η δυνατότητα του φάσματος και για την παρακολούθηση της κατάστασης ε, της ατμόσφαιρας ε, μέσω ειδικών διαστημικών εφαρμογών και στον τομέα των μεταφόρων. Εδώ έρχεται το σύστημα ε, GPS Γαλιλαίος όπως επίσης και άλλα έξυπνα συστήματα μεταφορών. Η επόμενη εγγεγραμμένη ομιλήθεια είναι η κυρία Νίμπλε, η οποία δεν φαίνεται στην αίθουσα. Και έτσι θα, το λόγο θα πάρει η κυρία Τόγια για 1,5 λεπτό παρακαλώ. κυρία Τόγια για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε μέχρι τώρα ότι μέσω αυτού του προγράμματος εναρμόνισης της αποτελεσματικότητα της σωστής χρήσης του φάσματος θα μπορέσουμε να επιβεβαιώσουμε μια διτή λειτουργία. Από τη μία θα πρέπει να απλοποιήσουμε την κατάσταση και από την άλλη να αναπτύξουμε το δυναμικό οικονομικής εκμετάλλευσης του συγκεκριμένου αυτού τομέα και για τις τηλεπικοινωνίες και για τα ραδιοτηλεοπτικά και για τις νέες υπηρεσίες δίδοντας μια νέα οικονομική όφηση σε όλους αυτούς τους τομείς ιδιαίτερα στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και εκμεταλλευόμενοι και τις πολιτιστικές και κοινωνικές δυνατότητες οι οποίες παρουσιάζονται. Κατά τη γνώμη μου, Επίτροπε, το πρόγραμμα αυτό θα πρέπει να είναι μια ευκαιρία έτσι ώστε οι επιλογές μας να επιβεβαιώσουν βασικές αρχές, πρώτη από αυτές τις αρχές, πλουραλισμό στα μέσα ενημέρωσης. Η αναθεώρηση του τρόπου κατανομής του φάσματος έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και θα πρέπει να οδηγήσει σε αποτροπή της συρροής ε, που, ε, φάσματος που δημιουργεί σε ολιγοπόλια και μονοπόλια που δυστυχώς σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες υπάρχουν και ενισχύονται. Δεύτερη βασική αρχή είναι η ισορροπία ανάμεσα στο άνοιγμα της αγοράς, τη φιλελευθεροποίηση της αγοράς, με τη δικαιοσύνη από την άλλη που επιτρέπει στην αγορά να προωθήσει και να υποστηρίξει και να διατηρήσει κάποιες ανηλυμένες υποχρεώσεις τις οποίες έχει αναλάβει στο παρελθόν. Τέλος, η διαφάνεια και η σωστή χρηστή διακυβέρνηση του φάσματος και της αδειοδότησης. Μιλάμε όχι μόνο για να αναπτύξουμε την αγορά η οποία θα πρέπει να υπακούει στις κοινωνικές ρυθμίσεις αλλά θα πρέπει επίσης να υπάρξει διασφάλιση ε, της εμπιστευτικότητας και σωστή χρήση των συχνοτήτων. Και αυτό είναι κάτι που δεν πρέπει να αγνοήσουμε για τις κοινωνικές πλευρές δεν έχω χρόνο. Αλλά παρόλα αυτά οι συνάδελφοι, οι προλελήσαντες αναφέρθηκαν και σε αυτόν τον τομέα. Για λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κυρία Κρός. Σήμερα γιορτάζει η Ευρώπη. Η Ευρώπη χρειάζεται απτά αποτελέσματα για τους πολίτες της. Ε, χρειάζεται μεγαλύτερη οικονομική ευρωστία, ευζήν για τους πολίτες της Ευρώπης. Ε, λοιπόν, η πρόταση του κυρίου Χόικμαρτ αντιστοιχεί πλήρως στις προσδοκίες των πολιτών διότι προσεγγίζει τους ε, πολίτες ε, στην Ένωση απελευθερώνει δηλαδή οι ζώνες ραδιοσυχνοτήτων για τις ασύρματες τεχνολογίες. Μέχρι το 2013 έχουμε θέσει προθεσμία για τα 800 MHz ε, και ε, για τα 1200 MHz 2015. Σωστές οι επιλογές μας αν θέλουμε να έχουμε τα πρωτεία στην Ευρώπη. 200 εκατομμύρια ευρώ είναι η αξία της νέας αγοράς. 3 έως 4% της οικονομικής ανάπτυξης εξαρτάται από, την, από τον τρόπο κατανομής των ραδιοσυχνοτήτων. Δείτε τα πρότυπα GSM που αποφασίστηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 90. εδώ μια σωστή όθηση στην οικονομία τη στιγμή που τη χρειαζόταν. Είναι σίγουρο ότι με τα νέα πρότυπα θα έχουμε κέρδος 80 Τις ε, δολάρια ε, ε, για κάποιες χώρες όπως η Ολλανδία που εκπρόσωπο έχουν προετοιμαστεί απελευθερώνοντας ήδη ραδιοσυχνότητες για την τέταρτη γενιά, το 4G. Για τους ραδιοκλητικούς δέκτες, για τις κρατικές εταιρείε, για θέματα παρεμβολών, για θέματα μικροφωνισμών θα πρέπει να βρούμε μία λύση. Ε, πρόκειται για τεχνικά ζητήματα που θα πρέπει να επιληθούν. Ε, και καλή τύχη πάντως ε, για να συνάψετε τελικά μια συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ κύριε συνάδελφε. Ο κύριο Ρούμπικ για δύο λεπτά θα πάρει το λόγο τώρα. Χωρί μικρόφωνο. Ναι, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα ζητώ συγγνώμη διότι έχουν εγκαταλείψει την αίθουσα μέλη, αλλά ψηφίζουν στην Επιτροπή, Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ήτρε και δεν μπορούν να, να απουσιάσουν από εκεί. Για τον συνάδελφο Χεκμάκ, Θέλω να πω ότι βρήκατε ένα καλό συμβιβασμό. Όμω σε αυτό το θέμα πρέπει πάντα να λαμβάνουμε υπόψη το επίπεδο δυναμικού και απόδοση που επιθυμούμε για το μέλλον. Αφενό για το, ε, το δίκτυο τέταρτη ε, γενεάς και από την άλλη πλευρά για του ε, καλωδιακού παρόχου και όσου συμμετέχουν όμως αυτό το επίπεδο απόδοσης ε, και επιδόσεων πρέπει να καθοριστεί. Πρόκειται πρώτον για τον όγκο στοιχείων και δεύτερον για τον χρόνο στον οποίο διαβιβάζονται αυτά τα στοιχεία, τα δεδομένα, ώστε να υπάρξει η συνύπαρξη των ε, διαφορετικών δυνατοτήτων και σε σχέση και με το λογισμικό software. Χρειαζόμαστε μια πιο εξειδικευμένη έκθεση για το μέλλον, ώστε το δίκτυο τέταρτης γενεάς ε, να μπορέσει να αυξήσει την ταχύτητά του όσοι συμμετέχουν μέχρι 100 megabits, megabytes είναι ε, σημαντικό αλλά πρέπει να αυξηθεί, αυξηθεί το δυναμικό. Εκεί όπου έχουμε μεγάλα προβλήματα είναι το επίπεδο τιμών ιδιαίτερα για την περιαγωγή, για το roaming. Υπάρχουν κράτη-μέλη που ε, για λιγότερο από ένα ευρώ αγοράζουν τέτοιες ε, δυνατότητες, εξαγοράζουν τέτοιες δυνατότητες τι γίνεται για το 9.900 ευρώ που κοστίζει σε μια χώρα και σε άλλη χώρα 14.900 ευρώ η ίδια ε, παροχή υπηρεσιών. Εδώ χρειαζόμαστε κατεπηγόντως επίτροπε να μεριμνήσουμε όχι μόνο το επίπεδο επιδόσεων να διασφαλίζεται σε αυτή τη νέα φάση αλλά και οι τιμές και να λάβουμε υπόψη το επίπεδο τιμών να έχουμε ένα κοινό επίπεδο, ενιαίο επίπεδο τιμών στην κοινή αγορά, κοινοτική αγορά, ώστε να μπορέσουμε να υποφεληθούμε των δυνατοτήτων. Εδώ έχουμε κατεπίγουσες προτεραιότητε που πρέπει να ανταποκριθούμε σε αυτές. Τώρα ερχόμαστε στη διαδικασία Catch the Eye. Ποιοι συνάδελφοι θέλουν να παρέμβουν. Έχει ζητήσει το λόγο ο κύριος Μόλζερ. Έχετε το λόγο για ένα λεπτό κύριε συνάδελφε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Ευρώπη μόνο για να προασπίσει αυτό το ρόλο του μεγαλύτερου ευρωπαϊκού χώρου έγινε ηγέτης της τεχνολογίας και η τεχνολογία αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική με τις νέες πολιτικές για το ραδιοφωνικό φάσμα θα πρέπει να προσπαθήσουμε να επιτύχουμε νέες ε, δυνατότητες ε, μετάδοσης. Και μια κεντρική ευρωπαϊκή διαχείριση δεν θεωρώ ότι είναι πολύ χρήσιμη. Ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηλώνει ότι θα μπορούσε να γίνει κάλλιστα σε εθνικά επίπεδο. Ένας ε, εθνικός ρυθμιστής δεν θα ήταν κακό και πέραν από το κόστο, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και το γεγονό ε, τη διάθεση περισσότερων δικτύων οπτικών ινών, διότι ακολουθούμε κατά πόδα ε, του οικονομικού μα ανταγωνιστέ, ε, ακόμα και την Κίνα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το ζήτημα αυτό συνεχίζει να παρακολύεται στη γραφειοκρατία. Θα πρέπει να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα για τι ραδιοφωνικέ συχνότητε. Τώρα το λόγο έχει η κυρία Κρόση, ε, Επίτροπος. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και όλους και όλες που συμμετέσχουν σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Φαίνεται πολύ τεχνικό το θέμα αλλά τελικά βλέπετε ότι είναι τόσο απλό σαν το αεράκι και το νεράκι. Όπως είπε και η Εκατερίνη Τράουτμαν, πρόκειται για δημόσιο αγαθό όσο και για εμπορικό. Και έρχομαι τώρα στον εισηγητή και τους κοιόδης που κατάφεραν το θέμα να το χειριστούν με τον ίδιο διαφανή και απλό τρόπο που απαιτείται. Σε μια δημοκρατία βέβαια χρειάζονται τέτοιες συζητήσεις. Κυρία Πρόεδρε, έχουμε ξανασυζητήσει το θέμα του ψηφιακού προγράμματος, συμφωνήσαμε όλοι ότι αν δεν αναλάβουμε όλοι τις ευθύνες μας και σαφή γραμμή, τότε μπορούμε και να ξεχάσουμε τι είχαμε προαποφασίσει ότι δηλαδή Πρέπει να ξέρουμε ότι μέχρι το 2020 και το γράφει αυτό στο πρόγραμμα πρέπει ένας Ευρωπαίος ή μία Ευρωπαία να μπορεί να πραγματοποιήσει ή να ανταποκριθεί στις ανάγκες του σε ψηφιακές συχνότητες. Κυρία Πρόεδρε, πρέπει λοιπόν να ρίξουμε κάποια συνέπεια για να καταφέρουμε τα, τους στόχους αυτούς. Ευχαριστώ όλους και όλες όσους και όσες μίλησαν γιατί τελικά πρέπει όλοι να συμφωνήσουμε στη στρατηγική μας προσέγγιση για διευθέτηση, διαχείριση του ψηφιακού φάσματος. Και αν μου το επιτρέπετε θα ήθελα να πω ότι έχω ένα θετικό προέστημα. Γνωρίζω ότι θα υπάρξουν εμπόδια, αλλά τα εμπόδια αυτά θα υπερπηδηθούν. Σεβόμαστε απόλυτα κυρία Πρόεδρε την χρήση του φάσματος για ψηφιακές δραστηριότητες, να μην υπάρξει εδώ καμία παρεξήγηση. Αφού μιλάμε για περισσότερες συχνότητες που πρέπει να διατεθούν για ευρυζωνική πρόσβαση, πρέπει να ξέρουμε επίσης ότι αργά ή γρήγορα και οι περισσότερες χώρες θα επιμένουν στο γρήγορα βέβαια πρέπει να εφαρμοστούν οι προτάσεις που κάναμε γιατί είναι κατάσταση γουίν-γουίν. Αν θέλουμε να δούμε να εμπνευστούμε από το παρελθόν, πράγμα που συνήθως δεν κάνουμε γιατί συνήθως εμπνευόμαστε από το μέλλον, τότε πρέπει να δούμε ότι σε σύγκριση με αυτά που ίσχυαν πριν από 15 χρόνια θα έπρεπε να πούμε ότι αν είχαμε τότε περιμείνει λέγοντας ότι πριν αποφασίσουμε οτιδήποτε πρέπει να είμαστε σίγουροι για όλα τότε δεν θα φτάναμε ούτε μέχρι τη σημερινή μας συζήτηση αν θέλουμε τη θέση 1 τη θέση 3 θα ήμασταν στην τελευταία θέση είναι βέβαια εθνική δικαιοδοσία το φάσμα, το γνωρίζω αυτό. Αλλά συμφωνούμε επίσης όλοι και όλες ότι το φάσμα είναι πολύ σημαντικός πόρος. Η ενιαία ψηφιακή αγορά είναι κάτι που σημαίνει ότι έχουμε και την ευθύνη και την ευκαιρία να δούμε τα πράγματα διαμεθοριακά και αυτό είναι κατεξοχήν διαμεθοριακό θέμα, τα φάσματα. Τώρα το χρονοδιάγραμμα και οι προθεσμίες. Είναι φανερό ότι το 2013 για μένα δεν είναι ημερομηνία πολύ βιαστική. Εμείς έχουμε κάνει τα πρώτα βήματα, πρέπει βέβαια να υπάρξουν συμφωνίες και με τις γειτονικές χώρες και αν τυχόν υπάρξουν απρόβλεπτες συνθήκες πρέπει και αυτές να βρούμε έναν τρόπο να τις αντιμετωπίσουμε αλλά χωρίς από διοπομπαίους τράγους και υπεκφυγές. Πρέπει να δράσουμε γρήγορα. Θα υπάρξουν λοιπόν εξαιρέσεις αλλά χωρίς καταχρήσεις τους. Και τελικά κυρία Πρόεδρε, προσβλέπω στην συζήτηση με το Συμβούλιο και στην, στα αποτελέσματα της ψηφοφορίας σας με εμπιστοσύνη δε προς το μέλλον. Οπότε και ένα από τα θεμέλια που έχουμε θέσει σήμερα θα έχει υλοποιηθεί πριν λήξει ο χρόνος. Σας ευχαριστώ ακόμη μια φορά για τις προσπάθειές σας, όχι μόνο τους ηγητές και τους κοιόδης, αλλά και όλους τους ευρωβουλευτάς των διαφόρων επιτροπών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κυρία Επίτροπε. Ο Κμαρος ηγητής μας θα κλείσει τη συζήτηση. Για δύο λεπτά έχετε το λόγο κύριε συνάδελφε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ κυρία Επίτροπε. Πρέπει να ξέρουμε ότι εδώ μιλάμε για πολύ ραγδαίες εξελίξεις. Ήταν ραγδαίες και θα παραμείνουν ραγδαίες. Ενώ πώς να προβλέψουμε λοιπόν το 2020 με τόσο ραγδαίες εξελίξεις. Όταν συζητούσαμε το θέμα των 700, τη συχνότητα των 700, Είχαμε πει ότι πρέπει αργότερα, αν χρειαστεί, να μπορέσουμε να προβλέψουμε εξαιρέσεις για να εκμεταλλευτούμε τις εξελίξεις. Διότι το φάσμα είναι δημόσιο αγαθό και πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε με όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερο τρόπο όπως είπε και η κυρία Τράουτμαν. Θα ήθελα όμως επίσης να τονίσω ότι δεν υπάρχει εδώ καμία διαμάχη μεταξύ εμπορικής και πολιτιστικής χρήσης. Θα ήθελα να καταφέρουμε να μπει και ο πολιτισμός μέσα σε αυτή την τεχνολογία, να μην περιοριστεί μόνο στην εμπορική χρήση. Αλλά αυτό θα γίνει αν δεν δείξουμε αρκετές φιλοδοξίες. Θα μείνει πίσω ο πολιτισμός που ήδη υστερεί στην Ευρώπη, υποφέρει. Νομίζω ότι μπορούμε να διασφαλίσουμε το συνδυασμό και νέων εμπορικών ευκαιριών και νέων πολιτιστικών ευκαιριών. Αλλά γι' αυτό χρειάζεται να μπορούμε να λαμβάνουμε αποφάσεις. Και το λέω χωρίς καμία ηρωνία ότι αλλά με μεγάλο βαθμό ικανοποίησης ότι κανείς εδώ σήμερα δεν αμφισβήτησε ότι πρέπει να είμαστε οι πρώτοι σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο. Ο ανταγωνισμός για τη γνώση σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε πρώτοι. Έληξε κυρίες και κύριοι συνάδελφοι η συζήτηση εδώ και η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Πέμπτη, την Τετάρτη, ε, συγγνώμη, μεθαύριο Τετάρτη στις 12.30 το μεσημέρι. Τώρα Ερχόμαστε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης